Και τώρα περνάμε στο πρόγραμμα εργασιών μας ε, με βάση το άρθρο 137 στις 12 Μαρτίου εγκρίθη το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης και διενεμήθη η ομάδα ΕΛΚ ζητεί δηλώσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νομική ασφάλεια των επενδύσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητεί να ε, συμπεριληφθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Μετά τις δηλώσεις αυτές θα ακολουθήσουν ε, οι ομιλίες ε, των μελών της ομάδας. Ο κύριος Ντόλ εξ του ΕΛΚ. Πρόεδρε, Ξέρετε τι συμβαίνει στην Αργεντινή υπό την ε, απειλή της εθνικοποίησης της εταιρείας ε, YPF όπου είναι ε, μέτοχος η Ρεψόλη, η Ισπανική εταιρεία. Ζητούμε να γίνει μια συζήτηση διότι όταν θέλουμε να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στις τρίτες χώρες πρέπει πάνω απ' όλα να αντιδράσουμε σε τέτοιες αυθαίρετες και μονομερείς ενέργειες όπως τη κυβέρνησης της Αργεντινής. Θα πρότεινα λοιπόν να γίνει μια συζήτηση αύριο να ε, καταρτιστεί και ένα ψήφισμα που δεν είναι ανάγκη να ψηφιστεί αύριο, θα μπορούσε να ψηφιστεί ίσως την Πέμπτη. Αυτό είναι το αίτημα της ομάδας μας. Ακούσατε την πρόταση του συναδέλφου Ντόλ. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης του συναδέλφου Ντόλ. Μισό λεπτό. Καταρχήν, βάσει του κανονισμού, πρέπει να ρωτήσω αν κάποιος θα μιλήσει υπέρ της πρότασης του κυρίου Ντόλ. Ο κύριος Μαγιώρο Ρέχα, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Μία αρχή που θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αρχή της ασφάλειας δικαίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε και να είμαστε εναντίον κάθε πράγματος που είναι αυθαίρετο εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ε, την νομιμότητά του. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια θέμητη ενέργεια που θα επηρεάσει εκατομμύρια μικρών μετόχων και που θα αποτελέσει ένα φοβερό προηγούμενο για τους Ευρωπαίους επενδυτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συζήτηση αυτή είναι εντελώς απαραίτητο να γίνει δεν μιλάω εδώ για τα συμφέροντα μιας ισπανικής εταιρεία. Ε, σκέφτομαι τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι ευρωπαϊκές εταιρείε από όλες τις χώρες μας, εκτός των συνόρων μας. Ε... Είστε λοιπόν υπέρ. Ε, ποιος είναι κατά της πρότασης. Κανείς. Ψηφίζομαι. Ποιος ε, συμφωνεί με την πρόταση του ΕΛΚ. να σηκώσει το χέρι παρακαλώ. Ψήφι κατά. Αποχές με κάποιες ε, αποχές έγινε δεκτή δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την ασφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ε, μπει στην ημερήσια διάταξη την Τετάρτη το απόγευμα για οι προθεσμίες Τετάρτη στις 12, αύριο 12 για, την, ε, για προτάσεις ψηφισμάτων. Ε, Κοινέ προτάσεις ψηφισμάτων έχουν προθεσμία στις 12 την Πέμπτη. Ε, ποιος θέλει να ε, ε, να υποβληθούν τροπολογίες. Ε, η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Παρασκευή στις 20. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μα για την απόφαση αυτή να οργανωθεί μια συζήτηση και να ε, προκύψει και ένα ψήφισμα. Όμω αύριο η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο δεν θα είναι εδώ, ε, διότι υπάρχουν κάποιες, ε, υπάρχει κάποια συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνα του ΝΑΤΟ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υποφεληθούμε από την παρουσία τη εδώ σήμερα για να μα κάνει μια σχετική δήλωση. με λίγο γιατί έχω ενημερωθεί ότι η ομάδα σας θέλει ένα ε, ειδικό σημείο στην ημερήσια διάταξη, το οποίο και αποφασίσαμε να το συμπεριλάβουμε. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση η πρόσθετη αυτή πρόταση. Ε, βέβαια, στις ε, παρεμβάσεις θα μπορέσετε πίσω αργότερα να επισέλθετε και στο ζήτημα αυτό. Τώρα, η έκθεση Λούλινγκ ε, για την φορολόγηση ηλεκτρικών ετών ε, ε, ε, ζητείται να αναβληθεί. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση Λούλινγκ, αλλά διατρέχει τον κίνδυνο να πέσει θύμα παρεξηγήσεων. Ε, πρόκειται για το ενεργειακό φορολογικό σύστημα, βενζίνη και ντίζελ, οικολογικά κριτήρια. Υπάρχουν φόβοι σε κάποιες χώρες ότι αυτή είναι μια έκθεση που σε τελευταία ανάλυση ε, θα καταστήσει ακριβότερα τα καύσιμα ιδιαίτερα για τα οχήματα ντίζελ. Ε, ιδιαίτερα τώρα που οι τιμές των καυσίμων είναι πολύ ψηλές ήδη. Διαπιστώνεται σωστά στην έκθεση και ότι αυτό θα γίνει αργότερα. Υπάρχει και μια διατύπωση όμως η οποία είναι κάπως αόριστη, ίσως είναι διατυπωμένη υπερβολικά αόριστη, ότι δηλαδή οι αυξήσεις τιμών θα αντισταθμιστούν στο, στην περίπτωση του ντίζελ. Όμως για το συμφέρον της έκθεσης και για χάρη της δικής μας οικολογικής συνείδησης, καλό είναι να αναβάλουμε την έκθεση και να διευκρινίσουμε τα θέματα που αφορούν το ντίζελ. Γι' αυτό υποβάλλω τη σχετική πρόταση. Είναι λίγο επιφυλακτική συνάδελφος Λούλινγκ, αλλά νομίζω ότι είναι και προς το συμφέρον της και προς το συμφέρον της έκθεσής της να υπάρξει κάποια διευκρίνηση με μια διατύπωση που αργότερα θα υποβάλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάμστορ θα μιλήσει για την ε, πρόταση. Στηρίζω την πρόταση να ε, φύγει η έκθεση αυτή από την τωρινή ημερήσια διάταξη. Χρειάζεται περισσότερη συζήτηση, όπως είναι διατυπωμένη τώρα ε, δείχνει ότι θα υπάρξει ακρίβεια και δεν θέλουμε να δώσουμε αυτό το πολιτικό μήνυμα. Χρειάζεται περισσότερη συζήτηση θέματα που δεν είναι επίμαχα μπορούν να προωθηθούν ε, στο Κοινοβούλιο με ταχύτερους ρυθμούς. Ποιος θέλει να μιλήσει κατά η κυρία Λούλινγκ. Θέλω να σας πω ότι δεν βλέπω κανέναν αντικειμενικό λόγο ε, να γίνει δεκτή, δεκτό αυτό το αίτημα της σοσιαλιστικής ομάδας. Ξέρετε κύριε Πρόεδρε, την περασμένη Κυριακή ο κύριος Σαρκοζή οργάνωσε μια συνάντηση στο, στην πλατεία Κονκόρντ και ε, ξεσήκωσε τα πλήθη λέγοντας «Μη φοβάστε». Όπως και ο κύριος Σαρκοζή, έτσι και εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι θα κερδίσω, αλλά ούτε και φοβάμαι. Εγώ πρέπει να σας πω ότι η διαβούλευση του Κοινοβουλίου πάνω σε αυτό το σχέδιο οδηγίας της Κομισιόν χρονολογείται από την 29η Απριλίου του 2011. Επί 7 μήνες συζητήσαμε το θέμα στην Επιτροπή. Η έκθεσή μου υιοθετήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου και έχουμε τώρα τέλη Απριλίου. Το να παρατείνουμε τις προθεσμίες δεν θα χρησιμεύσει σε τίποτα γιατί τα ζητήματα που διακυβεύονται είναι ξεκάθαρα. Ο κύριος Βόμποντα λέει ότι υπάρχει κάποια, υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Όχι. Και οι φιλελεύθεροι τάχθησαν σαφώς υπέρ της αύξησης και οι σοσιαλιστές το ίδιο όταν συζητήσαμε στην Επιτροπή. Εγώ ιτήθηκα στην Επιτροπή και υπάρχει η πρόταση να ψηφίσουν κατά γιατί στην αναλογικότητα αυτή. Όχι, ήθελα να το πω και στα γερμανικά για να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο των επιχειρημάτων των συναδέλφων. Αυτό το μήνυμα το πέρασαν στην Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, έρχεται μια στιγμή που δεν ε, μιλάει πια κανείς αλλά αποφασίζει και νομίζω ότι πρέπει να αποφασίσουμε αυτή την εβδομάδα. Κατανοητό, κυρία Λούλινγκ, δεν ήταν θέμα γλωσσικό αυτό. Ψηφίζομαι την πρόταση του συναδέλφου Σβόμποντα. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Α, νομίζω ότι θα πρέπει να ελέγξουμε. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Εψήφισαν όλοι, ξαναρωτώ. Μάλιστα. Πέρα τη ψηφοφορία λοιπόν. Απερίφθη η πρόταση αυτή. Η έκθεση λοιπόν παραμένει. Παραμένει η έκθεση στην ημερήσια διάταξη. Όχι, όχι κύριε Λάγκεν, σωστά τα λέμε. Τώρα, με βάση το άρθρο 90, πρόταση Γκουε για την συμφωνία με τη ΣΥΠΑ θα λάβει χώρα πριν από την ε, ψηφοφορία της έκθεσης της κυρίας για την έκθεση του κυρίου Κάτσμαρεκ για την διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας από την, ε, τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής. Προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών από τον εισηγητή και 76 μέλη και από εναλλακτικέ προτάσεις ε, ψηφισμάτων ε, είναι στις ε, Τετάρτη 18 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι. Αυτό είναι το πρόγραμμα των εργασιών. Περνούμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Χάουιτ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτών. Δίδω το λόγο καταρχήν στην ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κυρία Άστον. Λέβη Άστον.